Κυρίε Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ, ελάτε, ας καθίσουμε σιγά σιγά για να αρχίσουμε. Ελπίζω να χωρέσουμε όλοι, αν και δεν είμαι βέβαιος. Λοιπόν, όποιος βρίσκει να καθίσει, ας καθίσει. Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζω θερμά μαζί με την ε, Λίδια Γιαρόκα, τη Συμπρόεδρο, στην κοινή συνεδρίαση Επιτροπής Γυναικών και Νομικής Επιτροπής. Σήμερα θα ψηφίσω με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών συλλεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών και ερωτώ, υπάρχουν παρατηρήσεις από την πλευρά σας για την ημερήσια διάταξη. Βλέπω όχι. Είναι λοιπόν εγκεκριμένη. Η συμπρόεδρος επιθυμεί να μιλήσει και να πει κάτι ή μπορούμε να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ κύριε συμπρόεδρε. Είμαστε πολύ ευτυχής που συνεδριάζουμε μαζί σήμερα. Καλωσορίζω τους πάντες. Ε, λυπάμαι για την καθυστέρηση στην έναρξη. Υπήρχαν αλλαγές και στην αίθουσα και ήταν και μπλοκαρισμένα τα σανσέρ. Ελπίζω όλοι να πρόλαβαν και να πήγαν όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι η αίθουσα μας και συνήθως ε, γίνονται συνδιαλλαγές εδώ. Ελπίζω να μην χρειαστούν πολλές συνδιαλλαγές και να ψηφίσουμε εύκολα. Ανακοινώσεις του Προέδρου δεν υπάρχουν. Πάμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών από 9 Ιουλίου και 18 Σεπτεμβρίου. Αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής δεν υπάρξουν υποδείξεις για ε, τροποποιήσεις, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα και αυτά τα πρακτικά. Και τώρα πάμε στο σημείο 4 το καθοριστικό, η ψηφοφορία. Οι συνεισηγητές θέλουν το λόγο. Η κυρία ε, Κράτσα, η κυρία ε, Ρέγνερ, ποιος θέλει. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα πω μόνο ότι το θέμα αυτό προκαλεί πολλές συζητήσεις, είχαμε πολλές εντατικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις με τους σκιώδεις, τις σκιώδεις και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετασχόντες. Πάντοτε είναι επίπονη διαδικασία όταν οι συνεισηγητές καταπιάνονται με ένα θέμα. Εμείς στο πνεύμα της συνεργασίας προσπαθήσαμε παρά τις μεγάλες αντιθέσεις ε, μεταξύ μας να τα καταφέρουμε και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συνεργάτες μας από τις πολιτικές ομάδες και από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Κράτσα, δεν την βλέπω, τη συνάδελφο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή που οι δύο επιτροπές ε, θα ψηφίσουν ε, πάνω σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την οικονομία, την κοινωνία, το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως των γυναικών και πιστεύω ότι θα υποστηριχθούν οι συμβιβαστικές τροπολογίες και θα στείλουν ένα ηχηρό και συντεταγμένο μήνυμα για την δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Και προχωρούμε στην ψηφοφορία. Α, να διευκρινίσουμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Θα εφαρμόσουμε τη ε, διαδικασία της Νομικής Επιτροπής. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες με ε, ανάταση της χειρός. Αν, ε, τα, τις ε, αποχές θα τις λέμε. Αν θέλει κάποιος να γραφτεί η αποχή του να το πει. Ε, ηλεκτρονικά θα επαναλαμβάνουμε για έλεγχο, άμα δεν είναι σαφές. Και οι τελικές ψηφοφορίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες τις ηλεκτρονικές και να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και να ε? Δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα, με τη βοήθεια της γραμματείας θα καταμετρήσουμε αυτούς που δεν έχουν φέρει τις κάρτες. Τώρα, περνάμε στην ψηφοφορία και ψηφίζουμε κατευθείαν την τροπολογία 22 που είναι ταυτόσιμη με την 23. Υπέρ. Κάποιο ζητεί το λόγο, ψηφίζετε ή θέλετε να μιλήσετε. Α, θέλετε να ψηφίσετε. Η κυρία Κορνέλισεν. Διαδικαστικά. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει σήμερα να ψηφίσουμε για να προλάβουμε και να ολοκληρώσουμε πριν το τέλος της εντολής μας το θέμα αυτό. Όμως θέλω να επικρίνω λίγο τη διαδικασία, γιατί είχαμε μια συμβιβαστική συνάντηση και καθυστέρησαν πολύ συμβιβαστικές τροπολογίες. Η συνάντηση ήταν καλή οι εισηγητές είπαν ότι θα εξήταζαν μία σειρά από θέματα. Μετά οι συμβιβαστικές ήρθαν πριν από το Σαββατοκύριακο, χωρίς σχεδόν καθόλου αλλαγές. Και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για διαπραγματεύσεις ούτε για τίποτε. Οπότε ιδιαίτερα εμείς από τις μικρότερες ομάδες νιώθουμε λίγο ότι παραγωνιστήκαμε. Και τι χρειαζόταν η συνάντηση για τις συμβιβαστικέ αν δεν εγκρίθηκαν οι συμβιβαστικέ. Τέλος πάντων, επί της ουσίας ελπίζω να έχουμε καλό αποτέλεσμα, αλλά διαδικαστικά θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Εντάξει, λαμβάνουμε υπόψη μας την κριτική. Και τώρα 22 και 23 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκαν. Προχωρούμε 24 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Ε, έμπλενα Υπέρ. Ε, ε, έμπλενα ε, υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 171-72 μέχρι 190. Όλες θα τις ψηφίσουμε μαζί. Πέρα. Κατά. Απορρίφθηκαν. Συμβιβαστική Δύο. Υπέρ. Κατά. Αδεκτή. Τροπολογία 176 που φαίνεται... όχι πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε 176 πέρα. Κατά απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά δεκτή. ...186 υπέρ... ...κατά... ...απορρίφθηκε... ...συμβιβαστική 4 υπέρ κατά δεκτή. Λοιπόν, για να ξεφυλίσουμε λίγο εδώ, προσπερνάμε πολλά. Πάμε στη συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 6 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε την τροπολογία 6. Η συμβιβαστική τροπολογία 6. Σαράντα οχτώ 48 ψήφοι ήταν όλοι. 38 υπέρ, 9 κατά, καμία αποχή. Ωραία. Δεκτή όπως το είχαμε προείδη. ...291 της κυρίας Λούλινγκ, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 292 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 283, 93 ε, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 2,94 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 295 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 300 υπέρ. Κατά. Κάτι ξεχάσαμε. Α, ξεχάσαμε μία. 296. 296 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 300 υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε. Έλεγχος, έλεγχος. «26 υπέρ 22 κατά δεκτή». Ε, Έμπελ 58 υπέρ. Κατά. Και αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Την Έμπελ 58. «22 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται». Έμπελ 51 δεν θα την ψηφίσουμε. Τη τροπολογία 301 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 302 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. ΕΜΠΕΛ 59 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 55 υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός στην ΕΚΟΝ 55. Έντεκα υπέρ 36 κατά δύο αποχές απορρίπτεται. Έκον 56 υπέρ κατά Απορρίφθηκε. 303 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έλεγχος. 303. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. «28 υπέρ 19 κατά 3 αποχές δεκτή». «Εκον 57 υπέρ κατά Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Ο έλεγχος. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 57 ηλεκτρονικά. «28 υπέρ 21 κατά, δεκτή». Η 304 καταπίπτει. Πάμε στην 305 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλ 60 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 58 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 306 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 309 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπολ 61 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 59 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 312 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 313 έλεγχος. Ψηφίζουμε την 312 ηλεκτρονικά. «21 υπέρ 27 κατά δύο αποχές απορρίπτεται». «313 υπέρ κατά απορρίπτεται». Έκον 60 υπέρ κατά μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά αν θέλετε να κάνουμε έλεγχο θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την ΕΚΟΝ 60 ηλεκτρονικά. Δεκαεννέα υπέρ 28 κατά τρεις αποχές απορρίπτεται. Έμπουλ 62 υπέρ. Κατά. Έλεγχος Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την έμπλα 62. ...21 υπέρ 29 κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά δεκτή. 317 υπέρ κατά. Μα απορρίπτεται. 318 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Έμπλ 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλ 3 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλ 4 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλ 5 υπέρ. Κατά. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά να σιγουρευτούμε. Ναι. 21 υπέρ 28 κατά μία αποχή. 21 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Έμπλε υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την ε, έμπλεξη. Δεν ήταν σαφές σε το είδα εγώ. 38 προς 11. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 1 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 30. Εδώ έχουμε τμηματική. Πρώτο τμήμα. Περ. Κατά. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεκτό. Ήμκο 1 υπέρ. Κατά. Απεορίστηκε. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Προχωρούμε. 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. έμπλοχτο Α, έλεγχος. Την 38, μάλιστα, έλεγχος. Την 38. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέσσερις υπέρ 47 <laughs> κατά. Έμπλοχτό υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ένα. υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 39. Α, όχι, αυτή έχει τακτοποιηθεί. Πάμε στη 42 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έμπλε νέα τμηματική πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεκτό. Έκον 8 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έκον 9 υπέρ. Όχι, ε, την... Α, όχι, όχι, όχι, θα την ψηφίσουμε. Την έκον 9 θα την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έμπλ 10 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Α, εντάξει. Ε, σαφές έχει καταπέσει. Πάμε στη 46 υπέρ. Όχι, και αυτή είναι εντάξει. Ε, ναι, ναι. Πάμε στη 48. Ναι, ναι, τη λογική σκέψη 8, 48 υπέρ, κατά. Δεκτή. 49 υπέρ κατά απορρίφθηκε. έμπλα 11 υπέρ κατά δεκτή. Α, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την έμπλα 11. 28 υπέρ 24 κατά δεκτή. Έκον 10. Α, όχι, όχι, έχει καταπέσει. Τροπολογία 3, εντάξει και αυτό. Ήμκο 7, όχι, 50, 51, μάλιστα. Την 51 ε, της κυρίας Γιανακουδάκη, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 52, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 53, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Έκον 11 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ήμκο 8 τμηματική. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Θα έλεγα ότι είναι δεκτό, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της ΙΜΚΟ 8. 32 προς 17, τρεις αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Νομίζω ότι μάλλον απορρίφθηκε, αλλά για να δούμε. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε τη ΣΥΜΚΟ 8, το δεύτερο τμήμα. «27 προς 23 με δύο αποχές, δεκτό και αυτό». Τώρα, η 54 έχει καταπέσει, αν τα βλέπω καλά, 55 πρέπει να ψηφιστεί. Τροπολογία 55, υπέρ. Κατά. 55 υπέρ παρακαλώ άλλη μια φορά. Κατά. Μου φαίνεται ότι... Όχι, θα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί τα μπερδέψαμε. 29 προς 23 απορρίφθηκε. Δεκτή. Συγγνώμη, μπερδεύτηκε ο πρόεδρος. 29 προς 23 δεκτή. Η τροπολογία καλά που τα προσέχετε αυτά. 57 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά Δεκτή. Τι, δεν είναι, τι είναι, έχει καταπέσει. Το επόμενο, ΙΜΚΟ 10. Υπέρ, κατά, α, καφέ. Έκον 13, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός γιατί δεν ήταν σαφές. 13 προς 36 με τρεις αποχές απορρίφθηκε. Ήμκο 11 υπέρ. Κατά έλεγχος. Ήμκο 11 έλεγχος. «25 προς 23 με τρεις αποχές, δεκτή». «62 είναι ίδια με την ΕΚΟΝ 14, υπέρ» κατά δεκτές. Ήμκο 12 υπέρ κατά δεκτή. Ήμκο 13 υπέρ κατά έλεγχος. Την ε, Ήμκο 13 ηλεκτρονικά. 30 προς 21 με μία αποχή δεκτή. 63 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Έκον 15 τμήματική. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η 64 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 65 υπέρ. Κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 65. ...22 προς 28 με 2 αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 13 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 66 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Έμπλ 14 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, έλεγχος. Ψηφίζουμε την 68. 38 προς 12 με 2 αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ. Α, έχει καταπέσει. Ναι, ναι, ναι, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Πάει 4. Καταπίπτει. Προχωρούμε. Η 70 τώρα της κυρίας Λούλινγκ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έμπλ 15. Α, όχι, έχει καταπέσει και αυτή. 71, όχι, και αυτή έχει καταπέσει. Ε, 73 υπέρ. 73 υπέρ, κατά, δεκτή. Έκον 18 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά απορρίπτεται 74 υπέρ κατά απορρίπτεται Έμπουλ 16 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεκτό 5 υπέρ α όχι ε? είναι Εά, έχει καταπέσει. Ωραία, είναι σοφο, η σοφή γραμματεία. 41 υπέρ, κατά. Απερίφθη. Έκον 20 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Έκον 21 υπέρ, κατά. Να ψηφίσουμε τη 43. Όχι. Αφού. Όχι, λάθος ζητάει ο πρόεδρος. Τη 43 πρέπει να ψηφίσουμε το Χέκμαρ υπέρ. Αφού είπε η γραμματεία τη 43, δεν είναι ταυτόσιμη. Θα ψήφισουμε. τη 43. Έτσι κι αλλιώς θα απορριφθεί. Υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Έκον 21. Υπέρ, κατά, έλεγχος. Έκον 21. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 21 προς 28 μία αποχή απορριφθήκε. 77 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 86 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Ξεχάσαμε κάτι πάλι. Όχι, 87 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 89 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Το πρώτο τμήμα. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Της 92. «22 προς 29 απορρίπτεται». «93 υπέρ». «Κατά». Απορρίπτεται. «95 υπέρ». «Κατά». Δεκτό, δεκτή. Έκον 25. Υπέρ. Κατά. Όχι, έχει καταπέσει. Γιατί ψηφίσαμε την 95. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, σύμφωνοι. Προχωρούμε. 94 υπέρ. Όχι, όχι. Τόσο καλύτερο. Κατέπεσαν και αυτές. 102 τμηματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα. Αυτή δεν έχει καταπέσει. Κατά. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Ε, πέρα. Κατά. Δεκτό. Λοιπόν, δεκτό το δεύτερο τμήμα σε 102. Πάμε. Εκόν 27. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ε, την έκον 27 ψηφίζουμε. 22 προς 28 απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Μου φαίνεται ότι απερίφθη. Απορρίφθη. 106 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά απορρίπτεται έμπλ 21 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά έλεγχος τη τροπολογία 7 ηλεκτρονικά 32 προς 17 με 2 αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Η 9 θα ψηφιστεί ηλεκτρονικά. 38 προς 12, εντάξει, πέρασε. Μετά 107 υπέρ κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Τροπολογία 8 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 37 προς 13 με μία αποχή. Έμπλ 22. Α, όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει και δει κατά 10, 112. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 29. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 113 τροπολογία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 111 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν την ψηφίζουμε αυτή, έχει καταπέσει. Μάλιστα, μάλιστα, έχει δίκιο η γραμματεία. Εντάξει, και η 20 έχει καταπέσει, η ΜΚΟ 20. 115, ψηφίζουμε. Την... Ποιος είναι υπέρ της 115. Κατά. Απορρίφθηκε. Έκον 30 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 118. Όχι, εντάξει είναι αυτή. Πάμε στην 120. Την 120 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Ε, εντάξει, έγινε δεκτή. 123 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλ 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 122 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 32 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 125 υπέρ κατά απορρίπτεται 124 υπέρ κατά απορρίπτεται 127 27 υπέρ κατά απορρίπτεται 30α και 135 υπέρ κατά απορρίφθηκε 145 νίμπλερ υπέρ κατά απορρίπτεται 146 υπέρ κατά απορρίπτεται 147 υπέρ κατά απορρίπτεται 148 υπέρ κατά απορρίπτεται έκον 35 υπέρ κατά έλεγχος έκον 35 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε 26 προς 21 με 3 αποχές. Δεκτή 135. 149 έχει αποσυρθεί. 150 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 151 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Έμπλ 31 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 152 υπέρ. Κατά. Άλλη μια φορά. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίζουμε την 152 γιατί δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. «22 προς 28 με μία αποχή απορρίφθηκε». «158 υπέρ». Απορρίφθηκε. 160 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 157 υπέρ. Ε, έμπλ 33 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Έκον 37 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 159 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ε, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 159. 19 προς 30 με δύο αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλ 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 38. Υπέρ. Κατά. Α, δεκτή. Έκον 39. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Την ε, έκον 39 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 19 προς 30 απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, έλεγχος. 166 ψηφίζουμε. «21 προς 30 απορριφθήκε». Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Τη 12. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. ...37 προς 13, δεκτή. Τροπολογία 167 υπέρ. Κατά. Ε, δεκτή. Έκον 40 υπέρ. Όχι, καταπέσει. Ευχάριστο, να μην ψηφίζουμε κιόλα. Τώρα, η έκθεση συνολικά. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε όπως ήθιστε στη Συνομική Επιτροπή. Ε, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Εντάξει. 40 υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Τώρα θα ψηφίσουμε στο ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Πάλι ηλεκτρονικά. Το ίδιο αποτέλεσμα 40 υπέρ, 9 κατά, 2 αποχές. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για την απόφαση να γίνουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εδώ θέλω μυθική πλειοψηφία και εδώ ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. 41 υπέρ 9 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στις δύο εισηγήτριες και εύχομαι κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Καλώς. Πάμε στα, διάφορα, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Και μπορούμε εδώ να κλείσουμε την ε, συνεδρίαση.